kolegos, mes turime e, šiandienos komiteto e, vieną. Καλημέρα σα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση τη Επιτροπής μα. Έχουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε εδώ την κυρία Εντιτ Μπάουα που είναι εμπειρογνώμων από την ε, ΆΙΓΕ γιατί συνεργαζόμαστε με το ΆΙΓΕ και βεβαίως κυρίως με τους εμπειρογνώμονες. Λαμβάνετε σημαντικές αποφάσεις. Έχετε τη διερμηνία. Ωραία, πολύ ωραία. Η κυρία Μπάουερ λοιπόν ε, θα πάρει τώρα το λόγο, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Κάνει εισαγωγή, την ξέρουμε. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι και πάλι εδώ μαζί σας. Ήμουν μέλος της Επιτροπής για περίπου 10 χρόνια Τώρα είμαι μέλος ε, του Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων του ΕΙΓΕ. Εσείς με ορίσατε μέσω ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω αγγλικά. Γιατί έχω συντάξει ε, το σχέδιο της ομιλίας μου στα αγγλικά. Θα ασχοληθώ με τρία θέματα. Τι νέα έχουμε από, την, ε, από το έγε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων. Και επιπλέον ε, εκπονούμε την στρατηγική μας για τα επόμενα τρία χρόνια και θα ήθελα τη γνώμη σας για το πώς να διαμορφώσουμε την περαιτέρω εργασία μας. Είμαι η φωνή σας σε αυτό το φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Τώρα για το Ινστιτούτο το ίδιο. Εγώ υπερψήφισα τον κανονισμό εδώ στην Επιτροπή τη δική σας και φυσικά και στην Ολομέλεια για να δημιουργηθεί το Ινστιτούτο. Στην αρχή χρειάστηκε κάποιος χρόνος ε, και είχαμε πολλές δυσχέρειες. Μετά από τρία χρόνια επιτύχαμε να, επιτύχαμε να ξεκινήσει η πρόσληψη προσωπικού. Και χρειάστηκε να μετακομίσουμε. Ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή. Τώρα όμως πρέπει να σας πω ότι το Ινστιτούτο μας έχει σημειώσει μεγάλες πρόοδους, λειτουργεί κανονικά και έχει μεγάλο κύρος και σαφείς προοπτικές. Έχουμε παρκές προσωπικό, ε, βεβαίως ε, όχι ιδιαίτερα πολύ άριθμο. Το ΕΙΓΕ κάποτε το συνέκριναν με το ΦΡΑ ή το Eurofam, αλλά το ΕΓΚΕ πρέπει να σας πω ότι έχει ένα προσωπικό 50 υπαλλήλων, έχει επίσης μαθητευόμενους και αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Το Ινστιτούτο, ε, αυτό καθεαυτό έχει 37 υπαλλήλους προσωπικό. Το ΦΡΑ έχει άνω των 100 και το Eurofound ακόμη περισσότερους. 110, κάτι τέτοιο. Εάν ε, ε, επισκεφθείτε τον ιστοτόπο μας, θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Έχουμε επιγραμμικά επιγραμμικές εργαλειοθήκες για την ισότητα, για το δίκτυο ισότητας των φύλων. Ίσως αυτό η εργαλειοθήκη Συγγνώμη, καλύτερα ο δείκτης ίσως να είναι ο πιο ενδιαφέρον, το πιο ενδιαφέρον εργαλείο και θα ενημερωθεί τον προσεχή Οκτώβριο. Θα συμπεριλάβει και ένα νέο στοιχείο. Σε αυτό τον σύνθετο ενιαίο δείκτη αποφασίστηκε να συμπεριθούν στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών και δεν είναι εύκολο τώρα να ενταχθεί και αυτός ο δείκτης. Αυτό το στοιχείο στο δείκτη. Τώρα, να περάσω στο δεύτερο. Ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων επελέγει ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας που ασχολείται με τις στατιστικές φύλου και αυτόν το δείκτη ισότητας των φύλων. Σε μία από τις συνεδριάσεις μας πέρυσι Ασχοληθήκαμε σχεδόν αποκλειστικά με αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών γιατί παρουσιάζει δυσχέρειες. Ο δείκτης ε, περιλαμβάνει έξι στοιχεία με πολλούς υποτομείς. Τώρα δεν θα σας τα εξηγήσω, μάλλον ήδη τα ξέρετε και μπορείτε εύκολα και να τα βρείτε ε, στο site μας. Όμως για τη βία τίθενται πολλά θέματα. Γιατί έχουμε μόνο μία αξιόπιστη πηγή στοιχείων. Αυτή η έρευνα που έκανε πριν από μερικά χρόνια το ΦΡΑ. Δεν έχουμε τίποτα πιο πρόσφατο. Και ακόμη και τα στοιχεία από αυτή τη μελέτη και από την Eurostat γιατί και η Eurostat μας δίνει μερικά στοιχεία, αλλά είναι πολύ λίγα. Κυρίως για δολοφονίες, δολοφονίες κατά γυναικών, δολοφονίες γυναικών. Και δεν υπάρχει καν ε, εναρμονισμένος ορισμός για τα θέματα της βίας κατά των γυναικών. Άρα εδώ έχουμε δυσχέρειες. Αλλά συνεχίζουμε τη συζήτηση για το πώς θα ενημερώσουμε τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε και θέλουμε ιδιαίτερα να αποκτήσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Το άλλο θέμα που απασχόλησε το φόρουμ εμπειρογνωμόνων είναι οι τομές ανισοτήτων, εκεί που υπάρχουν επικαλυπτόμενες ανισότητες. Υπάρχουν μερικά μεθοδολογικά θέματα. Όπως ξέρετε είναι ένα στοιχείο κάπως παράπλευρο στο δίκτυ ισότητας των φίλων. Και το θέμα είναι μέχρι πού μπορείς να πας για να συλλέξεις στοιχεία για να εξακολουθήσουν να είναι αξιόπιστα. Γιατί υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς όπου επικαλύπτονται τα στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορούν να μπουν στο πεδίο εφαρμογής γιατί αλλιώ ακριβώς θα τα μετράγαμε δύο φορές. Φέτος προσπάθησαν να συμπεριλάβουν στοιχεία για τις αναπηρίες και την ηλικία και την ε, μεταναστευτική προέλευση. Το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων, όπως ξέρετε, είναι συμβουλευτικό σώμα του ΕΕΓΕ. Δυστυχώς δεν εκπροσωπούμεθα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΓΕ. Η επόμενη συνάντηση του φόρουμ αυτού θα γίνει αυτό το μήνα. Και γι' αυτό είναι σημαντική η ανταλλαγή απόψεων που έχουμε. Για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η στρατηγική μας. Και το τρίτο θέμα, ποια θα είναι η στρατηγική μας. Το ΕΙΚΕ έχει ήδη κάποιες ε, σκέψεις. Αλλά μέχρι να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά μπορεί να τροποποιηθεί οτιδήποτε. Το ΕΚΕ θα ήθελε να εργαστούμε προς τις εξής τρεις κατευθύνσεις. Το ένα θέμα είναι λοιπόν αυτός ο δείκτης ισότητας των φύλων, πρέπει να ενημερώνεται, πρέπει να εναρμονιστούν οι ορισμοί, και κάτι άλλο που θέλω να θέσω και εδώ για να με βοηθήσετε. Όπως ξέρετε, έχουμε, τίθεται το θέμα της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Μετά την επικύρωση από την Ένωση, θα υπάρξει υποχρέωση με βάση το άρθρο 11 αυτής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης να συλλέγουμε στοιχεία, να γίνουν έρευνες, ε, μελέτες για το θέμα αυτό. Οπότε θα χρειαστεί κάποιο συντονισμό. Και για το συντονισμό αυτό, στο καλύτερο πλαίσιο θα σημαίνει συμμετοχή της Επιτροπής του Κοινοβουλίου, της ΕΓΕ και ίσως και μη κυβερνητικών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο οργανωμένων. Για την εκτέλεση όμως, για την υλοποίηση του συντονισμού είμαι πεπισμένη ότι η είναι η έγκαια. Θα χρειαστεί όμως κάποια υποστήριξη στις προσπάθειές της αυτές. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να μας υποστηρίξετε στην κατεύθυνση αυτή. Αυτά όσον αφορά τον δίκτυο ισότητας. Ως ε, εκπρόσωπος αυτής της ομάδας εργασίας μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν γιατί οι ορισμοί εναρμόνισης ακόμη χρειάζονται ολοκλήρωση και βεβαίως έχει συντάξει ένα γλωσσάριο διαφόρων ε, ορισμών η ΑΕΚΕ. Θα, τον, ε, θα, τον βρείτε, θα το βρείτε και στο ιστότοπό της. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό τη ενσωμάτωση τη διάσταση του φύλου. Όπως σας είπα, είμαστε ένα σχετικά περιορισμένης έκτασης όργανο, άρα αναγκαστικά περιοριζόμαστε σε κάποια θέματα μόνο στη δουλειά που κάνουμε για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. στα δημοσιονομικά λοιπόν του φίλου περισσότερο και δει στο διαρθρωτικό και το επενδυτικό ταμείο εστιαζόμαστε στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσουν αυτά πολύ σαφή και σημαντική θεμενή αξία ως δουλειά της ΕΕΚΕ. Επιπλέον, και εδώ είναι το τρίτο στο οποίο προσπαθούμε να προχωρήσουμε, είναι αυτό το θέμα των γυναικών μεταναστριών. Θα χρειαστούμε όμως προσωπικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα των μεταναστριών. Ένα θέμα ασφάλειας πρωταρχικά και μια επιπλέον προσταμενή αξία που μπορεί να προσφέρει η ΑΕΓΕ με το έργο της. Αυτά για αρχή. Και θέλω να τι δικέ απόψεις γιατί είμαι η φωνή και τα αυτιά σα. Καλωσορίζω την ευκαιρία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε δυνατότητες για πιο τακτικές ανταλλαγές απόψεων αυτού του τύπου γιατί είμαι πεπισμένη πως είναι χρήσιμες για, σε, για σας όπως και για τις Αίγες. Ačiū, ponia eh, Edita Bauer. Iš tikrųjų, pritariu, kad eh, tas bendradarbiavimas ir keitimas. Σας ευχαριστούμε πολύ, Edita Bauer. Σίγουρα και εμείς eh, θεωρούμε αυτή τη συνεργασία ε, μεταξύ της Επιτροπής μας ε, και του ΕΓΕ εξαιρετικά σημαντική, σημαντική και για το Κοινοβούλιο αλλά και για την Επιτροπή μας. Αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα με την ε, ανταλλαγή απόψεών μας, κύριε Μούντι. Σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε σήμερα το πρωί εδώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καταρχήν θα ήθελα να αποτίσω, αν θέλετε, προτιμήσεις στο ΕΓΕ δηλαδή έχουμε ε, παρελειμμένα δει την ιστοσελίδα του ΕΚΙ, αλλά έχουμε συναντηθεί και με προσωπικό του ΕΚΙ και πραγματικά η υποστήριξή σας ε, ε, βρίσκει εκτίμηση από τη δική μα πλευρά και ο επαγγελματισμός σας. Επίσης, συμφωνώ με την τελευταία πρόταση που κάνατε ότι θα έπρεπε δηλαδή να ε, υπάρχει τακτική συμμετοχή του ΕΚΕ εδώ στις συνεδριάσεις μας για να μας ενημερώνει. Ε, είναι σημαντικό, ε, μεταξύ άλλων και για ένα από τα ζητήματα το οποίο αναφέρατε και το οποίο επιχαίρω ότι δείξατε, δηλαδή οι προπολογισμοί σε σχέση με τη διάσταση του φύλου, το gender budgeting, δηλαδή τόσο ο πρόεδρο όσο και άλλα μέλη εδώ τη Επιτροπή συμμετέχουν τόσο στην Επιτροπή Φύσκου όσο και στην Επιτροπή Προπολογισμών. Οπότε θέλουμε να ασκήσουμε περισσότερε πιέσει σε σχέση με αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια επίκυνται και σημαντικέ διαπραγματεύσει προπολογισμού. Θα ξεκινήσουν δηλαδή οι διαπραγματεύσει στο πλαίσιο τη ε, διάμεση ε, αναθεώρηση του Meeting Review που ε, βέβαια αποτελούν τα πρώτα βήματα προς το νέο πολιτευτές δημοσιονομικό ε, πρόγραμμα αλλά και τη διαμόρφωση των υπόλοιπων ε, προγραμμάτων, για παράδειγμα το πρόγραμμα πλαίσιο, το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο και άλλα. Ο προηγούμενος επίτροπος για θέματα προπολογισμού είχε αναλάβει είχε τη δέσμευση να υπάρξει αύξηση των σχετικών δαπανών για, τον, για τη διάσταση του φύλου στον προπολογισμό της Ένωσης. Ε, και θέλουμε να συνεχίσει η υποστήριξη του ΕΓΕ έτσι ώστε να παράγει δεδομένα που βασίζονται σε αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να αναπτυχθούν και τα εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν ακριβώς να προωθήσουμε την ε, συμπερίληψη ε, στην, ε, στους επροπλισμούς στη διάσταση του φύλου γιατί συχνά αυτά είναι τα μόνα δεδομένα τα οποία έχουν ακριβώς και μια τέτοια διάσταση του φύλου σε σύγκριση με τα εθνικά δεδομένα του κράτου μελών οπότε θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμο το να συνεργαστούμε στενά με το ΕΚΕ ειδικότερα ε, στο πλαίσιο των διάφορων επικείμενων οροσίμων αν θέλετε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκαρθία Περές. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας ε, καλωσορίζουμε εδώ, κυρία Μπάουερ. Κάτι τελευταία μας... Ε, Κάτι τελευταία μάλλον ε, ε, στη θητεία είχαμε ε, συνεργαστεί στενά και ε, ήταν πραγματικά πάντοτε πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία μας και εδώ στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής ΕΦΑΜ. Θεωρώ πως το έργο που επιτελείται στο ΕΚΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό και ο αντίκτυπός του. Αναφέρατε κάποια ζητήματα τα οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικά από την πλευρά του ΑΕΚ δηλαδή ισότιμη μεταχείριση, ε, το έργο που μπορεί να τελέσει το ΕΚΕ γενικότερα και ήδη αναφέρθηκε απανελειμμένα ότι θα πρέπει να υπάρχει τακτική ανταλλαγή απόψεων και να επιταθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και της Επιτροπής μας. Αυτό το έχω αναφέρει και εγώ και έχω αναφέρει επίσης ότι το έργο που επιτελεί το ΕΕΓΕ είναι χρήσιμο και για όλες εκείνες τις οργανώσεις και τα θεσμικά όργανα ε, τα οποία ακριβώς βασίζονται σε αυτά τα δεδομένα. Εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να έχουμε ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε ε, αυτά τα δεδομένα που παράγει το ΕΕΓΕ. Ίσως δηλαδή θα πρέπει να γίνουν κάποιες περαιτέρω προσπάθειες έτσι ώστε τα αποτελέσματα των εργασιών του ΕΓΕ να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται και ε, δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα της ισότητας ε, των φύλων. Κατά συνέπεια θα ήταν χρήσιμο να αυξηθεί και ο προπολογισμό ε, που προβλέπεται για το ΕΓΕ. Και εμείς θα ταχθούμε υπέρ αυτής της αύξησης και στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό. Δηλαδή, όχι μόνο θα πρέπει να παραμείνει στα επίπεδα του ο αλλά να αυξηθεί ακόμα περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις περαιτέρω αρμοδιότητες που αναλαμβάνει το ίδιο δηλαδή ε, συλλογή των δεδομένων, ανάλυση της σημερινής κατάστασης, αξιολόγηση βέλτιστων ε, πρακτικών και παραδειγμάτων ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εάν κάποια στιγμή έχετε οποιοδήποτε αίτημα από εμάς, από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών, για να σας βοηθήσουμε στην εργασία σας, βεβαίως ε, θα σας ακούσουμε. Βεβαίως να μας πείτε τι χρειάζεστε ως φορέας, θεσμικός φορέας της Ένωσης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υποφεληθούμε η μεν και η δε από την εργασία αντιστρόφως. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να λάβω το λόγο για το θέμα αυτό, ευχαριστώντας πρώτα την κυρία Edith Bauer για τη δουλειά της. Και έχω κάποιες ερωτήσεις. Εν γέννη μου φαίνεται πολύ καλή δουλειά του Ινστιτούτου για την ισότητα ευκαιριών και ο δείκτης νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί άπαξ και έχουμε ένα τέτοιο δείκτη μπορούμε να καταγράφουμε την κατάσταση σε διάφορους τομείς κοινωνικούς στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να πάρει περισσότερες αποχρώσεις αυτός ο δείκτης έτσι ώστε παραδείγματι να βλέπουμε και τις τάσεις αλλαγής, ε, την παρουσία γυναικών με αναπηρία, ε, προερχομένων από τη μετανάστευση κτλ. Ξέρω ότι είναι τετάνιο το έργο να δοθούν περισσότερες αποχρώσεις στο δίκτη. Εσείς ως ειδικό ασφαλώς έχετε πολλά ακόμα να προσφέρετε. Ερωτώ λοιπόν ε, τι ακόμα μπορούμε εμείς να σας προσφέρουμε ως υποστήριξη ώστε να ε, γίνει και πιο γνωστό στο κοινό το έργο του Ινστιτούτου. Γιατί βέβαια συναντούμε εκπροσώπους του Ινστιτούτου, κάνουμε προτάσεις για στρατηγικές επιλογές, κατευθύνσεις του Ινστιτούτου. αλλά θα ήταν καλό να καταστεί ευρύτερα γνωστό το έργο του. Για να μην ακούγονται όπως έχω ακούσει κάποιες φορές ρωτήσεις, μα χρειαζόμαστε ένα τέτοιο Ινστιτούτο. Θα πρέπει να σας γνωρίσετε δηλαδή περισσότερο ο κόσμος και οι ειδικοί να, ε, να αναγνωρίσουν την αξία του έργου σας. Τι λοιπόν άλλο θα μπορούσε να γίνει. Thank you really for, for your σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια. Τα σημείωσα και θα τα διαβιβάσω. Στο Διοικητικό Σύμβουλο του ΕΚΕ αλλά και του Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων τώρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα του προπολογισμού και την ε, λήψη υπόψη της διάστασης του φύλου εκεί. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη, ένα toolbox ε, σε ό,τι αφορά αυτό το ε, budgeting που έχει εκπονηθεί συλλογικά από το ίδιο. Είναι διαθέσιμη λοιπόν αυτή η εργαλειοθήκη, αυτό το toolbox και μπορεί ήδη να χρησιμοποιηθεί. Αυτό που μπορούμε εμείς να αναμένουμε είναι καθώς πρόκειται για ένα μικρό θεσμικό όργανο, είναι να θέτει μικρούς στόχους. Ε, και ε, σε αυτούς για τα επόμενα χρόνια ε, περιλαμβάνεται η καλύτερη αξιοποίηση, προσθέμενη δηλαδή αξία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διάστασης του φύλου από τα διαφορετικά ταμεία. Αυτό Πράγματι θα μπορούσε δηλαδή να αυξήσει τη χρησιμότητα του ΕΚΕ. Από εκεί και μετά δεν αποκλείουμε οι εργασίες μας να μπορούν να χρησιμεύσουν και για την λήψη υπόψη της διάστασης του φίλου στον προπολογισμό της Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ δηλαδή πως είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Θα είναι και κάτι νέο και θα έχει προσθέμενη αξία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κατά πόσο οι δείκτες ισότητας των φυλών αξιοποιούνται στο βαθμό που θα έπρεπε, η απάντησή μου είναι πως μάλλον όχι. έχουμε ε, λάβει πολλά αιτήματα συνεργασίας από την Επιτροπή και τα δεδομένα μας αξιοποιήθηκαν και από όλες τις προεδρίες του Συμβουλίου. Αποτελεί δηλαδή συνήθεια πρακτική το να επιλέγεται ε, ένας ε, ένα θέμα με αυτόν τον τομέα πάντοτε και ε, να αξιοποιείται στο πλαίσιο της κάθε Προεδρίας του Συμβουλίου. Όμως η συνεργασία, αν θέλετε, η αυτή αξιοποίηση των δεδομένων από το Συμβούλιο ε, δεν είναι τόσο ε, εντατική όσο από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Οπότε εκείνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι η δική σας Επιτροπή, εδώ θα μπορούσε να αξιοποιεί περισσότερο αυτά τα δεδομένα. Ορισμένες ε, δηλαδή φορές γίνονται αντιληπτά ως ε, ανταγωνιστικοί δείκτες αν θέλετε σε σχέση με εκείνους ε, του site της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά νομίζω πως για την Ευρώπη ο δικός μας δείκτης του ε πολύ ε, πιο κατάλληλος και μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ένα είδος βοηθητικού δίκτυου δημοκρατίας εντός ε, Ευρώπης. Για παράδειγμα, η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία εκπονείται ετησίως από την Επιτροπή Λίμπε, ε, υιοθετείται στη συνέχεια από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακριβώς ε, και ένα μια ενότητα σε ό,τι αφορά την ισότητα του και όπου ο συγκεκριμένο και οι συγκεκριμένοι δείκτε θα αξιοποιούνται πολύ συγκεκριμένα. Οπότε, σα καλώ να αξιοποιείτε σαν τα δεδομένα, ειδικότερα εδώ, στη δική σα επιτροπή, στι εκθέσει σα και από εκεί και μετά υπάρχουν και μια σειρά από περαιτέρω δυνατότητε υποστήριξη ε, την οποία μπορείτε να παρασχετε. Και θα πρέπει να σας πω ότι το Ε, γίνονται και από τη δική μας πλευρά ε, τέσσερα προσπάθειες ε, προς την ακριβώς καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων που παράγουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπάουερ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Θα συνεχιστεί και στο μέλλον ασφαλώς και περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις με ιδιαίτερη χαρά μας στηρίζουν πάντα στις εκθέσεις μας, στις νομοδοτήσεις μας, με τις, προ... με τις πληροφορίες που μας προσφέρουν. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη εντωμεταξύ και άρα δίνουμε ραντεβού.